Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχόλια σχετικά με τα υιοθετηθέντα, υιοθετηθέντα κείμενα και πρακτικά. Το επόμενο θέμα είναι οι συζητήσεις για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Η πρώτη συζήτηση αφορά τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και τους μαζικούς βιασμούς στην επαρχία του Νοτιού Κιβού. Μια στιγμή να βρω τον κατάλογο των ομιλητών. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο εισηγητή, τον κύριο Τάνοκ. Η λαϊκή δημοκρατία του ΚΟΓΟ δεν είναι πολύ δημοκρατία και δεν είναι και πολύ λειτουργική δημοκρατία αν είχε αναλάβει δράση η κυβέρνηση για να αποτρέψει αυτούς τους μαζικούς βιασμούς, δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεν έχει κάποιες δυνατότητες σε πάρα πολύ μεγάλα εδάφη της χώρας αυτής. Η βία είναι ένα ακόμη κεφάλαιο στην τραγική ιστορία αυτού του κράτους που οδεύει ταχύτατα στο να χαρακτηριστεί ένα αποτυχημένο κράτος. και μάλιστα ακόμα και όταν είναι γνωστοί οι δράστες των βιασμών ποτέ δεν θα δικαστούν. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας ε, κάνει να μην προσπαθήσουμε να ζητήσουμε να τιμωρηθούν. Νομίζω ότι υπάρχει δικαιοδοσία παγκόσμια στο ε, διεθνές εγκληματικό, στο διεθνές μάλλον ε, δικαστήριο, ποινικό και νομίζω ότι δεν μπορούμε σαν κοινοβούλιο να αγνοήσουμε αυτό το οποίο έχει συμβεί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ο επόμενος εισηγητής είναι ο κύριος Ρωμέβα Ρουέδα. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι με εντελώς διαφορετικό τρόπο για αυτό το οποίο συμβαίνει. Υπάρχει ένα ψήφισμα, το 1335, το οποίο υπογραμμίζει την ευθύνη όλων των κρατών να σταματήσει πλέον η ατιμορρησία και να διωχθούν όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας και ε, στην ε, σεξουαλική και άλλη βία εις βάρος κοριτσιών και γυναικών. Πρέπει να μην μείνουμε στην απλή καταδίκη και θα πρέπει και η κυβέρνηση του Κονγκό να αναλάβει τις ευθύνες της όπως και τα Ηνωμένα Έθνη και να τελειώνουμε με αυτές τις φρικαλαιότητες. Είναι απαραίτητο ε, να θεωρηθεί εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Ισλαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό η συγκεκριμένη καταπολέμηση της βίας της σεξουαλικής θα πρέπει να μην μένουν ατιμόρυτοι οι δράστες και θα πρέπει να ξεκινήσει η Εθνική Εκστρατεία Ενημέρωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φτάσει η ώρα να αναθεωρήσει τους όρους συνεργασίας με την χώρα αυτή που είχαν καθοριστεί στις αρχές του 2008 έτσι ώστε το θέμα καταπολέμησης των βιασμών να είναι ένας από τους βασικούς στόχους και θα πρέπει τα αναπτυξιακά ταμεία προς την λαϊκή δημοκρατία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως για να παρέχεται βοήθεια νομική και ιατρική στις γυναίκες και ε, στα κορίτσια που πέφτουν θύματα σεξουαλικής βίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια φορά ακόμη δυστυχώς το κοινοβούλιο μας πρέπει να καταδικάσει βία τις, ε, όλες αυτές τις εξάρσεις. Υπάρχει πρόβλημα με το μικρόφωνο σας. Μήπως μπορείτε να μετακινηθείτε. Τώρα με ακούτε, μάλιστα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μια φορά ακόμη το Κοινοβούλιο μας πρέπει να καταδικάσει ε, τις ε, βιαιότητες στην δημοκρατία του Κονγκό και ιδίως στο Νότιο Κιβού, διότι δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει επαρκής προστασία και πρέπει η κυβέρνηση ε, της χώρας να μπορέσει να προστατεύσει τα εδάφη και τους πολίτες, ιδίως τους, ε, ε, ε, τους αμάχους, διότι θα πρέπει μέσα στα πλαίσια αυτά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει τη χρηματοδότησή της διότι στο Νότιο Κιβού υπάρχει μία προτίμηση για την στρατιωτική λύση η οποία έχει αποτύχει και λυπούμεθα για την έλλειψη θάρρους της διεθνούς κοινότητος. Τέλος θα σας πω ότι και τα μέσα έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο τον οποίο δεν αναλαμβάνουν πάντοτε για να υπάρχει κινητοποίηση και για ενημερών με την κοινή γνώμη. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο επόμενος είναι ο κύριος Σάκε για ένα λεπτό. Η κυρία Σάκε. Ευχαριστώ η ευρεία τακτική των εναντίον των μάχων πρέπει ε, να σταματήσει και ε, να υπάρξει μια αναθεώρηση ε, της, των μεθόδων που χρησιμοποιούνται και ο ΙΕ έχει καταδικάσει τις εξάρσεις και πρέπει να σταματήσει η Πρέπει πρέπει να ε, ενημερώσουμε σχετικά με την σεξουαλική βία αλλά θα πρέπει να ε, καταδικάσουμε καταρχήν αυτές τις βιαιότητες. Οι γυναίκες ε, δεν ενημερώνουν διότι τότε τις αποκλείουν οι κοινότητές τους και θα πρέπει ποτέ να μην επιτρέψουμε να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις όπου εκατοντάδες χιλιάδες ατόμων, ιδίως γυναίκες υποφέρουν σιωπηλά. Υπάρχει ο ρηκτός πλούτος ο οποίος ούτως ή άλλως τροφοδοτεί ε, την διαμάχη στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ και τέλος η κυρία Ντεκάιζερ για 1,5 ε, λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε με μεγάλο θυμό και οργή ε, βλέπω να επανέρχεται αυτό το θέμα των ε, βιασμένων γυναικών ε, στο Νότιο Κιβού, στο Κόγκο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θα ήθελα μόνο να πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται τίποτα. Είπαμε για τη Μονούσκο, είπαμε για τον ΟΗΕ. Προετοιμάζεται νομοσχέδιο στο ίδιο το Κόγκο, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο για την δικαιοδοσία για τέτοιου είδους ε, αξιόπινες πράξεις. Σε αυτήν ε, την περιφέρεια της χώρας εξαναρχίζει ο πόλεμος, ε, προσοχή και υπάρχει και κάτι άλλο που δεν μπορώ να δικαιολογήσω με τίποτα. Ήρθαν οι γυναίκες εδώ στο κοινοβουλίο, τι ακούσαμε και ε, ούτε καν έχουν δικαίωμα για άμβλωση αυτές οι γυναίκες ε, που έχουν εμβιαστεί και τα παιδιά τους απορρίπτονται από όλε τις ε, κοινότητες. Είναι ένα δράμα και δεν θέλω να επαναφέρω μέσα στα καταπήγοντα το ζήτημα των εκτρώσεων. Απλώς η περίπτωση του βιασμού, ακόμη και όταν απαγορεύεται από το κείμενο δίκαιο η έκτρωση, αναγνωρίζει το δικαίωμα για έκτρωση όταν προέρχεται από το βιασμό. Και ε, σας λέω ότι αυτά τα παιδιά ε, απορρίπτονται από όλους στο Κονγκό. Πρόκειται για ένα ανθρώπινο δράμα και θα ήθελα να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το θέμα κάπου άλλο. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Σας ευχαριστούμε και τώρα από πλευράς ε, των πολιτικών ομάδων οι αγορητές ε, εκ μέρους του ΕΛΚΟ, κύριος ε, Κάσμαρικ, ένα λεπτό θα αρχίσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στο Νότιο Κιβού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η ένοπλη σύρεξη συνεχίζεται εδώ και χρόνια και καθημερινά υπάρχουν πράξεις βίας. Οι γιατροί χωρίς σύνορα εξ αρχής βοήθησαν πολλά θύματα βιασμού και συμφωνώ με την κυρία Ντεκάιζερ. Ε, είμαι και εγώ ε, απειδισμένος ε, με την κατάσταση γιατί αυξάνεται ο αριθμό των θυμάτων βιασμού στο Ανατολικό Κονγκό και γι' αυτό ξανασυζητάμε το θέμα. Αυτό πρέπει να κάνουμε όμω, γιατί η σεξουαλική βία είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεν μπορούμε να σιωπήσουμε ενώπιον των βιασμών. Δεν γίνονται πολλά από πλευρά ε, ε, του ΟΗΕ γιατί δεν υπάρχει καλή κατάρτιση, δεν έχουν ε, ούτε καν τα απαραίτητα όπλα. Αφήστε που υπάλληλοι και ανώκρανοι ορισμένε φορέ βιάζουν αυτέ τι γυναίκε ε, εμείς συνταπανίσαμε 7.000 ευρώ για να παρακολουθήσουμε τις εκλογές στον Κογκόμα. Ας δώσουμε αυτά τα λεφτά για να γίνουν οι προσφυγές ενώπιον της δικαιοσύνης για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό η κυρία Γκόμες τώρα. Η σεξουαλική βία στο νότιο Κιβού πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνα και πρέπει να ε, τιμωρηθούν οι δράστες ούτω ώστε στο μέλλον να αποφύγουμε τέτοιες αποτρόπες πράξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναδείξει σε προτεραιότητα αυτό το θέμα στα πλαίσια της συνεργασίας της ε, με το Κόγκο και να δακτυλοδεικτήσει για αυτές τις επιχειρήσεις ε, που για να εκμεταλλευτούν τον ορεκτό πλούτο υποστηρίζουν τις ένοπλες ομάδες, ε, τις παραστρατιωτικές ομάδες που εμπλέκονται σε αυτές τις πράξεις βίας. Θα πρέπει Επίση, να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν ναι, ε, και άλλε απαράδεκτε πράξει. Ο Αγκουστίνο Σεγκάη, για παραδείγματο χάρη, ε, στι 22 Ιουνίου συνελήφθη στο αεροδρόμιο ε, του Κονγκό, ερχόμενο από την Αγγόλα. Και πώ έγινε αυτό, βάσει ενό μαύρου καταλόγου των αρχών τη Αγγόλα, που όμως όμω αρνούνται αυτό το αίτημα κράτηση αυτού του ανθρώπου. Παραβιάζονται καθημερινά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και αμέσω πρέπει να απελευθερωθεί ο Σεγκάγια και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει σε αυτό. Ευχαριστούμε από πλευρά των φιλελευθέρων η κυρία Μπιλμπάου. Ένα λεπτό. Για μια ακόμη φορά οι γυναίκε είναι τα θύματα αυτή τη υπόθεση. Αυτών των πολεμικών σειράξεων μάλλον. στην ουσία η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται σαν όπλο καταστροφής. <clears throat> Μην ξεχνάμε επίσης και τα οικονομικά συμφέροντα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο δραστηροί στον εμπορικό τομέα, στον τομέα της εκμετάλλευσης των ορυκτών καρπών του πολέμου αυτού. Νομίζω ότι θα πετύχουμε περισσότερα. Πρέπει να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος, θα πρέπει να στηρίξουμε τη δημοκρατία στο Κονγκό. Ο μόνος τρόπος είναι αυτός για να αποτρέψουμε τη γενικευμένη σύραξη. Πρέπει να υποστηρίξουμε την πολιτική διαδικασία γιατί μόνο έτσι θα αποφύγουμε, όπως είπα, την πολεμική σύραξη. Τσαρνέσκι, ένα λεπτό. Είμαστε λίγοι σήμερα το απόγευμα εδώ, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε εδώ και να μιλάμε και μιλάμε στο όνομα της Ευρώπης. Υπάρχει αναρχία πολύ μεγάλη σε αυτή τη χώρα δυστυχώς. Οι αρχές όμως δεν είναι ανίσχυρες. Έχουν κάποια μορφή εξουσίας, έχουν την αστυνομία, έχουν στρατιωτικούς οι οποίοι δυστυχώς όμως λειτουργούν με αυθαίρετο τρόπο και δεν βοηθούν συστηματικά τα θύματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ασχολείται με το θέμα αυτό για πρώτη φορά, δυστυχώς. Για μια ακόμη φορά απευθύνουμε μια έκκληση λοιπόν στην κυβέρνηση της λαϊκής δημοκρατίας έτσι ώστε να προσπαθήσει επιτέλους να προστατεύσει τις γυναίκες πολίτες. Όπως είπε και ο κύριος Κάτσμαρεκ, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε να δούμε πώς δαπανώνται τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου στη χώρα αυτή. Ο κύριος Μπέλτερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχα μια τηλεφωνική επαφή με ένα Ολλανδό που εργάζεται στο Ανατολικό Κονγκό στο Κιβού σε μια φιλανθρωπική οργάνωση. Είναι ιδιαίτερα ευτυχής που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται σήμερα με αυτή την τραγωδία την οποία βιώνει ο πληθυσμός του Κονγκό. Πρόθεσή μας είναι να καταδικάσουμε αλλά όχι μόνο τις φεκαλαιότητες και την άκρατη αυτή μορφή βίας. Θα πρέπει να δούμε και ποιος είναι ο ρόλος της Μονούσκο, της ενοπλής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών και πώς μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά σπάζοντας έτσι αυτήν την πυκνή αίσθηση σιωπή η οποία συνήθως χαρακτηρίζει τα θύματα αυτής της σύραξης. Δυστυχώς οι έρευνες που είχαν ξεκινήσει για τα θέματα αυτά δεν έχουν ακόμα οδηγηθεί σε θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Όμπερ Μάιερ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο ο Κονγκό έχουν μία παράδοση πεντηκονταετίας και ε, από την εποχή που ήταν ε, ε, βελγική απικία και ήταν υποχρεωτική καταναγκαστική εργασία για τον πληθυσμό. Θα πρέπει κάθε φορά που δεν ε, εκπληρωνόντουσαν οι στόχοι να τιμωρεί το, ο πληθυσμός και νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να επανορθώσει τα, τις αδικίες τις οποίες έκανε. Βλέπουμε όμως τώρα νέα βία με εμπόλεμες καταστάσεις όπου ο κάθε φύλαρχος θέλει να αποδείξει τη δύναμή του και να καταστρέψει και ε, ε, εκτός από τις γυναίκες τις οποίες επιτίθενται καταστρέφουν και όλες τις οικογένειες και μετά ε, το επόμενο είναι ότι ε, οι οικογένειες αυτές καταστρέφονται σε, στη δημοκρατική λοιπόν δημοκρατία του Κονγκό θα έπρεπε να προσαχθούν ή στα δικαστήρια οι υπέτη αλλά στις λίγες περιπτώσεις όταν οι γυναίκες ε, καταφεύγουν στα δικαστήρια υπάρχει προστασία για αυτές αλλά θα μπορούσαμε να εξασκήσουμε οικονομική πίεση διότι δεν είναι δυνατόν να ζητούμε τα πλούτη του Κονγκό και από την άλλη πλευρά ε, να καλύπτουμε τους εγκληματίες. Αυτή ήταν, ε, αυτή ήταν η λίστα των ομιλητών και τώρα μεμονωμένα οι επόμενοι ομιλητές και, με καταρχήν την κυρία Μακαβόη. Ευχαριστώ. Ε, η κατάσταση στην ε, ε, επαρχία του Νότιου Κιβού βλέπουμε ότι κάθε μέρα υπάρχουν 40 βιασμοί από στρατιώτες ή από προσκύμενους στο στρατό. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια ούτε ιατρική, ούτε ηθική, ούτε πολιτική και πρέπει να προστατεύσουμε τα θύματα. Μέχρι στιγμής έχουμε 170 θύματα και μάρτυρες οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μια ανεξάρτητη ε, ε, ε, έρευνα κατά τρόπον ώστε να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι έκαναν τις διάφορες πράξεις αυτές τον Ιούνιο για να καταδικάσουμε την, την, ε, ε, την κατάσταση. Ο κύριος Παλέξης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Η βία η οποία σοβεί στη χώρα αυτή τροφοδοτείται από την έλλειψη ατιμορρησίας και δυστυχώς διαδίδεται σαν επιδημία και φοβάμαι ότι και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο διεθνές δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Η ατιμορρησία αυτή ισχύει από ό,τι φαίνεται και για τους ίδιους τους εκπροσώπους της ένοπλης ε, δύναμης των Ηνωμένων Εθνών εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσει να βρει κάποιους άλλους τρόπους για να βοηθήσει τα θύματα και τις οικογένειές τους και θα πρέπει επίσης και κάποια διεθνή βιομηχανικά μονοπόλια που εκμεταλλεύονται τις πρώτες ύλε της χώρας αυτής να μην το κάνουν εις βάρος του φτωχού εργατικού δυναμικού. Θα πρέπει να βοηθήσουν και αυτοί. Ο κύριος Κέλλιν. Είναι τραγική ιστορία αυτή για, το, για τη λαϊκή δημοκρατία του Κογκό, Όσα ακούσαμε μέχρι τώρα είναι δυστυχώς κάτι το οποίο ευτυχώς έχουμε σταματήσει να ακούμε εδώ και καιρό. Υπάρχει βέβαια το θέμα της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της συγκεκριμένης χώρας που κανονικά θα έπρεπε να βοηθούν τη χώρα αυτή να πλουτίσει αλλά υπάρχει βέβαια και το θέμα της τραγικής θέσης στην οποία βρίσκονται ε, οι γυναίκες και τα παιδιά της χώρας αυτής. Άνω των 70 γυναικών βιάστηκαν και αυτό είναι υπερβολικά σοβαρό σαν θέμα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να υπάρξει μια κάποια λογική αλλαγή στην κατάσταση και θα πρέπει να είναι δυνατή η κυβέρνηση εκεί έτσι ώστε να καταπολεμήσει την ατιμορρησία και να αποδώσει δικαιοσύνη. Ευχαριστώ η κυρία Κρέτου για ένα λεπτό. Δεν είναι η πρώτη φορά όπου συζητούμε για την κατάσταση στη λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο. Δεν καταδικάζουμε μόνο τις φρικαλαιότητες ε, αλλά και επίσης καταδικάζουμε την αδράνεια της κυβέρνησης της κεντρικής της χώρας. 12 στρατιωτικοί μόνο προσήχθησαν στη δικαιοσύνη ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 400.000 ε, λέει η ομιλήτρια γυναίκες που έπεσαν θύματα βιασμού. 48 ε, γυναίκες πέφτουν θύματα βιασμού αναώρα στην λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Οι βιασμοί είναι ταμπού εν τω μεταξύ και οι γυναίκες αυτές αποκλείονται από τις οικογένειές τους, απομονώνονται από την κοινωνία και νομίζω ότι πρέπει πλέον κάτι να κάνουμε. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στρέψει επιτέλους την προσοχή της, τουλάχιστον σε ιατρικό και σε κοινωνικό επίπεδο για τις γυναίκες αυτές και να υπάρξει ένα ειδικό διεθνές δικαστήριο για την ε, δημοκρατία του Κονγκό. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ζητήσω από τους Ευρωπαίους πολιτικούς να δώσουν κάρτες παραμονής στα θύματα βιασμού που πρέπει να μπορούν να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώπη. Και τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye και πρέπει να σας πω ότι έχω περισσότερες αιτήσει από ό,τι φοβάμαι ότι θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε. Αλλά αν περιορίσετε το χρόνο ομιλία σας θα δούμε πώς θα πάμε. Η κυρία Εσάγια καταρχάς. Ευχαριστώ. Ε, το Ανατολικό Κομβό υπάρχει αστάθεια και εδώ και χρόνια και η σεξουαλική βία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά. Ε, χιλιάδες γυναίκες έχουν βιαστεί και ο αριθμός αυξάνεται συνέχεια σύμφωνα με τις ε, διεθνείς μαρτυρίες και επίσης υπάρχει έρευνα διότι φαίνεται ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι καταγράφεται στις στατιστικές του ΟΗΕ. Ε, υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις και έξω στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίοι πρέπει ε, να ε, επιβληθούν στο Κονγκό για να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι με την βοήθεια του ΟΗΕ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο Κονγκό υπάρχει μια σειρά περιπτώσεων ξεκάθαρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να τις καταδικάσουμε. Ε, οι βιασμοί κυρίως βέβαια στρέφονται εις βάρος των γυναικών και αυτό το οποίο χειροτερεύει την κατάσταση είναι ότι οι δράστες, οι βιαστές πολλές φορές είναι μέλη του, ε, ε, του στρατού της χώρας. Μιλάμε για μαζικούς βιασμούς και μάλιστα τα θύματα όχι μόνο υφίστανται αυτή την απαράδεκτη βία αλλά πολλές φορές απομονώνονται από την κοινωνία τους και πολλές φορές καταλήγουν σε μη επιθυμητές ε, γεννήσεις. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τουλάχιστον τον στιγματισμό των θυμάτων. Θα πρέπει τα θύματα να τύχουν μιας κάποιας ψυχολογικής τουλάχιστον βοήθειας. Πρέπει να καταδικάσουμε όλους αυτούς τους βιασμούς με οποιαδήποτε μορφή διεξάγονται και θα πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας αυτής για να σταματήσουν οι απαράδεκτες αυτές καταστάσεις. Αυτή η μαζική βιασμοί στο Κονγκό είναι κάτι το οποίο μας κάνει να αγανακτούμε. Αλλά δυστυχώς τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχουν τόσες πολλές ε, μορφές βίας στη χώρα αυτή, περισσότερα θύματα από ό,τι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν ήδη οι Κογκολέζοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να δείξει αλληλεγγύη, να απαιτήσει να τιμωρηθούν οι βιαστές και να βρεθεί μια δύσκολη λύση σε μια απαράδεκτη κατάσταση. Αυτά όλα όμως θα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να δώσουμε μια γρήγορη οικονομική βοήθεια για να καταπολεμήσουμε τη σεξουαλική βία και να βοηθήσουμε τα θύματα. Βασική μας προτεραιότητα είναι η ιατρική βοήθεια. Δεν μπορούμε να δώσουμε ιατρική βοήθεια αν δεν έχουμε χρήματα. Πρέπει να βοηθήσουμε επίσης την κοινωνική επανένταξη των θυμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, δύο φορές στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχαμε εκπροσώπηση τις ε, επαρχίες του Κιβού και μας είπαν τι γίνεται αλλά και τι κάνουν οι ίδιοι για να μπορέσει κανείς ε, να ε, συλλάβει και να φέρει στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους. Μας είπαν όμως ότι τον τελευταίο χρόνο δεν ήταν δυνατόν οι εκπρόσωποι του, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Κονγκό να συναντήσουν αυτές τις γυναίκες και ε, να μάθουν τι έχει γίνει. Αντιθέτως μας είπαν ότι αντετάθησαν όλες οι προσπάθειες. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει να ε, επανορθώσει την κατάσταση γιατί δεν είναι δυνατόν τα προγράμματα τα οποία αποβλέπουν στη βοήθεια των θυμάτων να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν. Η κυρία Κόχολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. αυτό που συμβαίνει στο Νότιο Κιβού σε στρατιωτικό επίπεδο οδηγεί σε αυτά τα κρούσματα, τους βιασμούς που ταυτόχρονα υπάρχει ε, η υπερβολική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας ε, και συγκεκριμένα αυτής της περιοχής. Αλλά ε, το βασικό είναι να προστατεύσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά γιατί χρησιμοποιεί το βιασμός ως όπλο και εδώ μιλάμε για γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού και στη συνέχεια αποξενώνονται και απομακρύνονται από τις κοινότητές τους. Πρέπει να βρούμε μία λύση, πρέπει να αντιδράσουμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ πρέπει να αναλάβουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα, ούτως ώστε να ε, σταματήσουν αυτοί οι βιασμοί στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και το Κονγκό πρέπει να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια της ε, βοήθειας που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των γυναικών και των παιδιών και όχι για κάτι άλλο. Πρέπει να σταματήσουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να βάλουμε ένα τέλος και στη διαφθορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εφόσον ε, υπάρχει ένα σύστημα και ε, δεν έχουν προσταχθεί στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι χαιρετίζω την παράταση της θητείας του κλιμακίου του ΟΗΕ και θεωρώ ότι θα πρέπει να φροντίσουμε η εντολή αυτή να εφαρμόζεται και σωστά να μην βιάζονται οι γυναίκες να μην ε, υφίστανται τις οικονομικές επιπτώσεις όλες οι οικογένειες και να ληφθούν ψηφίσματα και μέτρα ε, που καταδικάζουν ε, διεθνώς αυτές τις πράξεις. Πώς μπορούμε όμως να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση μέχρι το 2003 όπου πέθαναν και σκοτώθηκαν 5,5 εκατομμύρια άτομα και πρέπει να συμβάλλουμε στο να υπάρξει επίλυση του θέματος. Ευχαριστούμε η κυρία Ρόη ε, ε, πρόκειται για τις χειρότερες μορφές ταπείνωσης αυτές που βιώνουν οι γυναίκες ε, στο Κόγκο. Απομονώνονται διαβίου από την κοινότητα οι γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού και επικρατεί η ατιμορρησία για τους στρατιώτες και για τους παραστρατιωτικούς. Η παράταση της εντολής των δυνάμεων του ΟΗΕ είναι απαραίτητη αλλά δεν επαρκεί για την προστασία των πολιτών. Ο πρόεδρος Καμπίλα δήλωσε ότι θα ακολουθήσει η προσέγγιση μηδενικής ανοχής για τους βιασμούς και θα ερευνήσει το θέμα. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται πρόγραμμα επανένταξη ε, στην κοινωνία. Χρειάζονται κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση συγκεκριμένο νόμο για να απογορευτεί η εκμετάλλευση των ορεικτών στο νότιο Κιβού. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, λέει η κυρία Πλάμπε, φυσικά έχω ε, μελετήσει τα έγγραφα που καταγράφουν τον αριθμό των θυμάτων βιασμού στο Κονγκό, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε η κυρία Ντεκάιζερ. Πήγε επί τόπου και είδε με τα μάτια της ε, ε, το τι υποφέρουν οι γυναίκες, τον τρόμο στα μάτια τους και στα μάτια των παιδιών τους. Θα πρέπει να ζητήσουμε ρητά να σταματήσει αυτό, να κινηθεί το Κοινοβούλιο, όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, οι αρχές ε, του Κονγκό πρέπει να διερευνήσουν τις υποθέσεις αυτές ε, και να διώξουν τους υπετίους και ταυτόχρονα εξασφαλίσουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη για όλα τα θύματα που θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα προστασίας. Η διεθνής κοινότητα, όλες οι διεθνείς οργανώσεις για την περάψη των δικαιωμάτων πρέπει να εμπλακούν για να σταματήσει αυτή η κατάσταση στο Κονγκό. Και τέλος ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτοί οι μαζικοί βιασμοί συνεχίζονται εδώ και δεκαετίες. Θα πρέπει λοιπόν η δράση μας να είναι ισχυρή. Πρέπει να βοηθήσουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που βοηθούν τα θύματα. Πρέπει να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια νομοθετική πρόταση αντίστοιχη με την πράξη του Αμερικανικού Κογκρέσου που επιβάλλει περιορισμούς στην χρήση των πρώτων υλών που προέρχονται από τη χώρα αυτή, έτσι ώστε αυτοί που ανέχονται τέτοιες ενέργειες να είναι υπόλογοι για τις πράξεις τους. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβουμε δράση. Τώρα στρέφομαι στην Επίτροπο, κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές για την προσέγγιση την οποία είχαν. Φυσικά ε, όλοι είδαμε τα τρομακτικά αυτά νέα από το Κιβού όπου μια ομάδα ενόπλων επιτέθηκαν και βίασαν μεγάλο αριθμό γυναικών με συστηματικό τρόπο. Αυτοί οι εγκληματίες... Φαίνεται ότι ήταν οι μάγοι μάγοι που αποστάτησαν από τον στρατό του Κονγκό ε, επειδή δεν κατάφεραν να ενταχθούν σε αυτόν μετά από πολύ καιρό. Ε, είναι απαράδεκτα αυτά τα εγκλήματα και φυσικά νιώθουμε όλοι μεγάλη ανησυχία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε τα γεγονότα και ε, να διώξουμε τους δράστες. Μας ενημέρωσαν ότι ο Γενικός Εισαγγελέα της Λαϊκής Δημοκρατίας ε, του Κονγκό ε, με την υποστήριξη της Μονούσκο θα μεταβεί επί τόπου για να συλλέξει νομικά ε, τεκμήρια και να προετοιμάσει τη δίωξη. Ζητούμε από τις αρχές ε, της λαϊκής δημοκρατίας ε, του Κονγκό να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με αυτό το θέμα και να απονείμουν δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά, τον δηλώνουμε απειβισμένοι δεν επαρκεί και το αντιλαμβάνομαι κι εγώ, οπότε όλοι μας θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες δράσεις θα πρέπει να αναλάβουμε και μέσα από το ε, Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη Μονούσκο. Υποστήριξη προς τα θύματα. Φυσικά αυτό πρέπει να είναι η άμεση προτεραιότητα της Ένωσης, η οποία ήδη έχει αναλάβει δέσμευση για παροχή ιατρικής περίθαλψης, ε, για την ε, ελάφρυνση του πόνου των θυμάτων. Ε, ε, χρειάζεται λοιπόν κατά προτεραιότητα η ιατρική περίθαλψη. Αυτή είναι μια συμπεφωνημένη προτεραιότητα εδώ στην Ένωση και σα ενημερώνω ότι είμαστε ε, στο μέτωπο ε, και υποστηρίζουμε όχι μόνο αυτό και δράση για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή αυτή. Επίσης ενημερωτικές εκστρατείες, ασκούμε πολιτική πίεση. Όλα αυτά είναι επιμέρους στοιχεία της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Η σεξουαλική βία και ο βιασμός εξαπλώνονται στη λαϊκή ε, Δημοκρατία του Κόγκο. Το 2009 σημειώθηκαν πάνω από 15.000 κρούσματα, 15.000 βιασμοί. Αυτό ανέφερε ο ΙΕ για το 2009. Οπότε πρέπει να επιτεθούμε στη ρίζα του κακού και να μεριμνήσουμε ώστε η δικαιοσύνη του Κονγκό να μην έχει μόνο περιστασιακές και σπασμωδικές αντιδράσεις. Στο Στην ανατολική περιφέρεια του Κόγκο δεν υπάρχει κράτος δικαίου διότι ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί ποιος κατέχει την εξουσία. Η σεξουαλική βία συνεχίζεται και διαιωνεί στην υποδέστερη θέση που κατέχουν οι γυναίκες ολόκληρη τη χώρα. Αυτό έχει ιδιαίτερα αντικό αντίκτυπο προς ε, τα παιδιά που θα γεννηθούν λόγω αυτών των βιασμών, όπως μας είπε η κυρία Ντεκάιζερ. Για να βελτιωθεί η κατάσταση θα πρέπει να συνεχίσουμε και στρατιωτική και μη στρατιωτική δράση κατά ε, των επαναστατών και από αυτήν την άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι τέτοιου είδους σειράξεις σε πάρα πολλές φορές όπου εμπλέκονται ομάδες που δεν έχουν όμως σαφή πολιτικό προσανατολισμό ή όπου εμπλέκονται εγκληματίες από γειτονικέ χώρες είναι ένα θέμα που δύσκολα μπορεί μπορούμε να Παρόλα αυτά είναι ολένα και πιο επίγον να κάνουμε αποφασιστικά ε, μέτρα για να δώσουμε μια απάντηση η δικαιοσύνη, η αστυνομία, η άμυνα, ο στρατός του Κονγκό δεν είναι στο ύψο των περιστάσεων. Αυτό μας ανησυχεί και γι' αυτό ε, καλούμε τις αρχές ε, του Κονγκό να αποδώσουν και πάλι μέγιστη προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Εάν δεν σημειωθεί ουσιαστική Πρόοδο ε, στον τομέα της δικαιοσύνης και της άμυνας ε, θα τεθεί να αμφιβόλει πρόοδος ε, που έχει σημειωθεί στον τομέα της κοινωνίας, της οικονομίας κτλ. Και επειδή επίκυνται εκλογές νομίζουμε ότι πρέπει όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις του Κονγκό να εμπλακούν ενεργότερα διότι το μέλλον της χώρας διακυβεύεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη παρέχει υποστήριξη για τη μεταρρύθμιση του τομέα της στο πλαίσιο των κοινών αποστολών της ΚΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς ε, και υπάρχει και η διμερής υποστήριξη από πλευρά των κρατών μελών. Αυτές οι δράσεις εστιάζονται στην ανάγκη καταπολέμησης σεξουαλικής βίας και παραδείγματος χάρη η Europol έστειλε μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα ε, σεξουαλικής ε, βίας στην Κόμα. Είναι μια πόλη στο νότιο Κιβού. Επίσης ε, πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ψυχολογικά τα θύματα. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα αν βρούμε ένα κοινό έδαφος συνεργασίας με τα κράτη-μέλη αφενός και με τις κογκολέζικες αρχές αφετέρου. Ε, πλην όμως σε αυτό το τομέα η ίστατη ευθύνη ούτως ή άλλως θα είναι στα χέρια της ίδιας της λαϊκής δημοκρατίας ε, του Κονγκό και η κυβέρνηση πρέπει να δείξει πραγματική αποφασιστικότητα και να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Ευχαριστώ. Έχω λάβει ε, έξι προτάσεις ψηφισμάτων για να λήξει συζήτηση. Λίγη συζήτηση και θα ψηφίσουμε ε, τα ψηφίσματα μετά τις επόμενες συζητήσεις. Περνάμε τώρα στην Ινδονησία συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον μειονοτήτων